από ένα στοιχείο το οποίο αναφέρατε εσείς ε, προηγουμένως σε σχέση με το ρόλο του Κοινοβουλίου. Εσείς ε, το αποκαλέσατε ε, επίκεντρο, καρδιά της δημοκρατίας. Εμείς δεν έχουμε εδώ συστήματα για να λειτουργήσουν τα πράγματα, αλλά τα πράγματα λειτουργούν μονάχα εάν όλοι σέβονται το σύστημα. Εσείς μιλήσατε για ισότητα φύλων, μιλήσατε για την μεγάλη σημασία που έχει το γεγονός που ίσως μια γυναίκα θα είναι για πρώτη φορά πρόεδρος της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά συνέβησαν και χτες ε, ε, εδώ στην Ολομέλεια ε, που ε, δεν ψηφίστηκε. Μία γυναίκα από την Πολωνία η οποία δεν ψηφίστηκε ε, πρόεδρος στην Επιτροπή Απασχόλησης εδώ στο ίδιο το Κοινοβούλιο για λόγους τελείως διαφορετικούς από τους κανόνες που πρέπει όλοι να σεβόμαστε. Χωρίς σεβασμό των κανόνων δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε. Di ή θα πρέπει να συνενέσουμε όλοι ε, να βασιστούμε στον κανόνα ντεχόντ ή διαφορετικά δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε. Ε, και γιατί εσείς ε, θα σκεφτείτε περισσότερο τα θέματα αυτά. Εσείς γράψατε κάποιες επιστολές και ξέρετε όμως ότι τα λόγια είναι επεαπτερόεντα ενώ μονάχα τα γραπτά παραμένουν. Εσείς γράψατε και στην ομάδα Ρινιού και στους σοσιαλιστές επίσης. Γι' αυτό ζητούμε εμείς κάποιες διευκρινήσεις όπως άλλωστε ζήτησαν διευκρινήσει και άλλε ομάδε. Ε, σε σχέση, α πούμε, με αυτά που είπε η συνάδελφο Γκαρσία ε, Πέρε, ε, τι σα ρώτησε. Σα ζήτησε διευκρίνηση όσον αφορά τον μηχανισμό του κράτου δικαίου. Εμεί, λοιπόν, θέλουμε να ξεκαθαρίσετε πραγματικά το θέμα αυτό στην απάντησή σα, αλλά βεβαίω εμεί έχουμε τελείω εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη, γιατί αν μιλάμε για αυτή την μεταετή περίοδο, τότε εμεί βρισκόμαστε στην εντελώ αντίπερα όχθη. Επομένω, χρειάζεται οπωσδήποτε διευκρίνηση όσον αφορά αυτό το μηχανισμό για το κράτο δικαίου. Επίση, θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο αντιμετωπίζουμε την κλιματική αλλαγή, γιατί επί τη κλιματική αλλαγή μπορεί να υπάρχουν πολύ θετικά θέματα. Ναι, τα αναφέρατε. Ε, αυτό το Just Transition Found ας πούμε, αυτό το, ε, ε, αυτή η τράπεζα για τις βιώσιμες επενδύσεις, όλα αυτά πάρα πολύ καλά. Αλλά εδώ στην ουσία προσπαθούμε να υψώσουμε διαρκώς το ύψος των φιλοδοξιών μας, χωρίς όμως να λέμε με ποιο συγκεκριμένο τρόπο θα επιτύχουμε αυτές τις υψηλότατες φιλοδοξίες. Χρειαζόμαστε διευκρινήσεις, γιατί όλα βρίσκονται σε μια γενική ασάφεια. Ε, όσον αφορά τους κλιματικούς στόχους, ήταν 50% την προηγούμενη εβδομάδα, 55% τώρα. Ε, δεν το καταλαβαίνουμε ε, ε, εδώ. ακούσαμε περισσότερο δηλώσεις προθέσεων παρά συγκεκριμένες, συγκεκριμένα θέματα. Και επίσης το θέμα της κοινωνικής πολιτικής. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα βεβαίως και είναι ένα θέμα ε, το, στο οποίο στάθηκε πάντα με επικριτική στάση η ομάδα μας γιατί ε, αυτή ε, η ελάχιστη αμοιβή που θα διασφαλίσει το ελάχιστο εισόδημα των νέων ναι αλλά με ποιους πόρους πρέπει να μας τα πείτε αυτά. Επίσης όσον αφορά την μετανάστευση σήμερα το πρωί μας δώσατε ένα δείγμα γραφής εξαιρετικό αλλά ήταν στην ουσία ένα σχολικό παράδειγμα. Μας είπατε για αυτόν τον Σύρο πρόσφυγα, στον οποίο ανοίξατε την αγκαλιά σα στη Γερμανία και έμαθε γερμανικά. Αλλά κοιτάξτε, ε, όλοι, ε, οι δεν είναι πρόσφυγε, υπάρχουν μετανάστες. Ε, υπάρχουν μετανάστε οι οποίοι είναι απολύτω παράτυποι μετανάστες. Και από την δική μα άποψη όλα αυτά τα οποία συνέβησαν και την προηγούμενη εβδομάδα είναι εξαιρετικά σημαντικά. Δηλαδή ένα άνθρωπο, ένα άτομο το οποίο βρίσκεται υποδικαστική διερεύνηση στη χώρα μας γιατί έχει παραβιάσει του τους ναυτικούς κανόνες της Ιταλίας ε, αποτελεί αντικείμενο συζήτησης στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και μάλιστα μπορεί να προκύψει και κάποια ακρόαση όσον αφορά το θέμα αυτό. Εκεί θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις γιατί βάσει αυτών των απαντήσεων θα μπορέσουμε και εμείς με μεγαλύτερη ευκολία να λάβουμε απόφαση ε, μετά το πέρας των συζητήσεών μας. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Σίντερμαν. Έχετε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Φοντελάιν. Ε, έγινε λόγος για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ε, κατά κόρον έγινε λόγος για αυτούς ε, και τις τελευταίες ημέρες έχω πάρει χιλιάδες ηλεκτρονικά μηνύματα και ίσως και άλλοι συνάδελφοι που έχουν ως αντικείμενο την υποψηφιότητά σας. Και θέλω λοιπόν να δράξω την ευκαιρία να παραθέσω κάτι από αυτά τα μηνύματα. Εκεί αναφέρεται το εξή και παραθέτω. Ως ψηφοφόρος πιστεύω και ελπίζω ότι ε, θα έχουμε μία γυναίκα που θα εκλεγεί πρόεδρος επιτροπής ε, και η κυρία που στέλνει το μήνυμα Αναφέρει επίσης όμως ότι δυστυχώς το να εκλεγεί μια γυναίκα η οποία υπήρξε υπουργό Άμυνα, αυτό σημαίνει στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης. Τέλος της παράθεσης. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ στη συνάντηση που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ήρθατε σε εμά, τη δική μας την πολιτική ομάδα και μας παρουσιάσετε το δικό σας το όραμα για το μέλλον της Ευρώπης. Κατέστησα σαφές ότι το δικό μας το όραμα είναι τελείως διαφορετικό. Και να σας εξηγήσω εμείς είμαστε η μόνη πολιτική ομάδα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που απορρίπτουμε κατηγορηματικά τη συνέχιση της πολιτικής λιτότητας. Εσείς μιλάτε για το μέλλον της Ευρώπης και θεωρώ ότι πρέπει επιτέλους να ε, έρθετε σε ρήξη με αυτή τη νεοφιλελεύθερη πολιτική. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή η πολιτική λιτότητα δεν οδήγησε σε εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών, οδήγησε στο αντίθετο. Τι έγινε, είχαμε έλλειψη επενδύσεων στην παιδεία, στην υγεία και επίσης ε, δεν υπήρχαν πλέον πόροι έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το, η κλιματική αλλαγή. Αυτοί που υπέφεραν από αυτή την πολιτική λιτότητα ήταν οι πολίτες ε, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η κυρία Φοντελάιν, όποιος θέλει να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή πρέπει να δράσει τώρα, χωρίς καθυστέρηση. Όποιος θέλει να αντιμετωπίσει την, ε, τις υποδομές πρέπει τώρα να επενδύσει και όποιος επιθυμεί την κοινωνική ασφάλεια στην Ευρώπη πρέπει όπως σας είπα να έρθει σε ρήξη αυτή τη στιγμή με την πολιτική λιτότητα. 113 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε φτώχεια ή απειλούνται από τη φτώχεια. Περιμένω λοιπόν από μια υποψήφια για τη θέση της Προέδρου να μην λέει μόνο ευχάριστα λόγια, ε, να πει ξεκάθαρα ότι χρειαζόμαστε μια κοινωνική επίθεση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πει ότι εγώ θέλω σε πέντε χρόνια κανένας Ευρωπαίος πολίτης, ανεξάρτητα που βρίσκεται, σε ποια περιφέρεια, να μην απειλείται από τη φτώχεια και να μπορεί να διάγει έναν αξιοπρεπή βίο. Για να γίνουν όμως αυτά πρέπει να υπάρχουν οικονομικές προϋποθέσεις. Αλλά στο θέμα της φορολογικής πολιτικής σήμερα παραμείνατε πολύ γενικοί. Αυτά τα βελούδινα γάντια που χρησιμοποίησατε δεν είναι το σωστό εργαλείο για να έχουμε μια αποτελεσματική πολιτική. Εγώ θέλω λοιπόν μια υποψήφια να είναι ε, αποφασιστική, να έρθει σε ρήξη με του ομίλου επιχείρησεων, να πει εγώ θα σπάσω το dumping το φορολογικό, θα κλείσουν οι φορολογικοί παράδεισοι. Επιτέλου ε, θα υπάρχει μια δίκαιη φορολογική πολιτική, επιτέλου θα υπάρχει δίκαιη φορολόγηση. Και Επίσης, ε, να επενθυμίσω ότι υπάρχουν και αυτά τα δισεκατομμύρια ε, που θα επενδυθούν σε ευρωπαϊκούς εξοπλισμούς. Το είπατε εσείς αυτό, αλλά αυτά είναι χρήματα που θα έπρεπε να επενδυθούν στην υγεία και στην παιδεία. Ε, δεν θα επενδυθούν όμως εκεί, αλλά θα επενδυθούν σε σύγχρονα οπλικά συστήματα. Και μάλιστα σήμερα, σήμερα κάποιοι ονειρεύονται και ένα στρατό στο διάστημα. Για μας αυτό είναι φιάλτης, δεν είναι όνειρο. Το να μιλάτε εσείς ε, για ευρωπαϊκό στρατό, ο στόχος είναι απόλυτα σαφής. Να υπάρξει επανεξοπλισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στρατιωτικοποίηση της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς ως αριστεροί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το απορρίπτουμε κατηγορηματικά. Ε, θέλουμε οι διενέξεις να επιλύονται με διαφορετικό τρόπο, να υπάρχει για μας, ας πούμε, είναι απαραίτητος απαραίτητο να υπάρξει μια διάσκεψη για τον αφοπλισμό. Τελευταίο μου θέμα, τα ευρωπαϊκά εξωτερικά σύνορα αυτή τη στιγμή είναι τα πιο θανατηφόρα του κόσμου. Και θεωρώ ότι είναι δήλωση χρεοκοπία τη Ευρωπαϊκή πολιτική, το ότι κάθε μέρα πεθαίνουν άνθρωποι στη Μεσόγειο, ενώ εκείνοι που υπερασπίζονται τα οικουμενικά δικαιώματα, ε, πολλοί εξ αυτών ποινικοποιούνται. Και άκουσα τι είπατε κυρία Φαντελάιν. εμεί ε, ω αριστεροί θα είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά την εφαρμογή τη πολιτική σα. Το δικό μα το πρόγραμμα για το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια κοινωνική Ευρώπη, Ευρώπη με αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αυτά που είπατε εσείς δεν έχουν καμία σχέση με το δικό μας το όραμα και γι' αυτό το λόγο και εμείς δυστυχώς θα σας καταψηφίσουμε. Ο κύριος Φαράζ έχει το λόγο εκ μέρους των μη εγγεγραμμένων. Για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Όπως ε, σας είπα και την τελευταία φορά, δεν θα με χάσετε, να εδώ θα ήμουν και να εδώ είμαι. Το ευρωπαϊκό, το δικό μας το κόμμα, τα πήγε πάρα πολύ καλά στις εκλογές, κερδίσαμε πάρα πολλούς. Επανήλθα λοιπόν σε ένα χώρο ο οποίος έχει ταπεινωθεί. Ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέστησε αυτό το χώρο αδρανή ε, και σήμερα υποτίθεται, σας δίνεται κάποια δύναμη, μπορείτε να την αδράξετε. Είδατε, ο κύριε Φαντελάν σήμερα είναι μια προσπάθεια της Ευρωπαϊκής να προσπαθήσει να ελέγξει ακόμα και το τελευταίο κομμάτι της ζωής μας. Θέλει να έχει μια συγκεντρωτική, μη δημοκρατική Ευρώπη, ένα είδος κομμουνισμού θέλει η κυρία Φοντελάιεν. ένα είδος κομμουνισμού όπου το κράτος θα ελέγχει τα πάντα, όπου ε, τα εθνικά κοινοβούλια θα πάψουν να παίζουν οποιοδήποτε ρόλο. Και να σας πω ε, αυτό που αφορά εμάς. Ε, πρέπει να σας πω, δεν μας χαλάει αυτό, κάπου μας αρέσει κιόλα. Γιατί με τον τρόπο αυτό, ξέρετε τι κάνετε, κατορθώνετε να φτιάξετε το Brexit ακόμα πιο δημοφιλές στην Αγγλία. Δόξα το Θεό. Όσον αφορά όμως ε, την άμυνα, η κυρία Φοντελάνη είναι φανατική. Θέλει να έχει ευρωπαϊκό στρατό. Όμως δεν είναι μόνη της και όταν υπάρξει αυτός ο ευρωπαϊκός στρατός πάρα πολλά πράγματα θα χαθούν στην Ευρώπη. Ο κύριος Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος, την Κυριακή, την ημέρα της Βαστίλης, μπήκε σε ένα ανοιχτό αυτοκίνητο με όλες αυτές τις δυνάμεις, τις στρατιωτικές πίσω του, κοιτάζοντας τον κόσμο με τη μορφή ενός νέου επικαιροποιημένου Ναπολέοντα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Πέντε χρόνια με τέτοιους ανθρώπους μετά από πέντε χρόνια η Ευρωπαϊκή Αμυντική Άμυνα θα έχει ολοκληρωθεί. Και αυτό όμως που χρησιμοποιείται για την άμυνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την επίθεση. Και εμείς ως Κοινοβούλιο δεν θα μπορούμε να ελέγξουμε τίποτα. Γι' αυτό καταψηφίστε την. Ψηφίστε υπέρ της δημοκρατίας. Ψηφίστε υπέρ των πολιτών σας. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Φάρατζ. Και Τώρα θα ακούσουμε την απάντηση της ε, κυρίας Φόντε Λάιεν. Θα απαντήσει στις παρεμβάσεις των αρχηγών των πολιτικών ομάδων. Παρακαλώ κύριε Φόντε Λάιεν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να σας πω τελείως ειλικρινά, ακούγοντας τον τελευταίο μιλητή, ε, νιώθω πάρα πολύ καλά. Καταλαβαίνω το πόσο πολλοί οι Βρετανοί θέλουν ε, να συνεργαστούν ε, μαζί μας, αλλά ευτυχώς ε, υπάρχετε κι εσείς από τους οποίους πολύ ευχάριστα θα παρετηθούμε και θα απομακρυνθούμε. Και ακριβώς αυτό είναι το ωραίο σε αυτή την Ευρώπη. Σε αυτή την Ευρώπη βλέπουμε ότι υπάρχουν κράτη τα οποία έχουν έρθει ε, με τη δική τους βούληση. Κανείς δεν τα ανάγκασε. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι από κοινού, ότι ενωμένοι είμαστε πιο ισχυροί, μπορούμε να προσπιστούμε αξίες που είναι σημαντικές για μας. Γνωρίζουμε ότι τα καθήκοντα που επίκυνται στον στον κόσμο είναι τόσο μεγάλα που κανείς από εμάς δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει μόνος του. Όμως, αν συνεργαστούμε, αν αναπτύξουμε μία δύναμη, μία ήπια δύναμη, ε, θα είναι μια καθαρά ευρωπαϊκή δύναμη που θα βασίζεται στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είναι μια δύναμη που θα μας κάνει δυνατούς, που θα μας δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το μέλλον, να μπορέσουν τα παιδιά μας να προχωρήσουν με πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Και τώρα λοιπόν θα μπω σε ορισμένα συγκεκριμένα θέματα. Κοινωνική οικονομία της αγοράς. Ε, πρόκειται για κάτι το καθαρά ευρωπαϊκό και έχουμε αυτή την θαυμάσια σύνδεση ανάμεσα σε μια εύρωστη οικονομία με άλλου κοινωνικού παράγοντε. Γνωρίζουμε όμω ότι όλοι μα μπορούμε να εργαστούμε σε αυτή την εύρωστη οικονομία. Αυτό λοιπόν το παράδειγμα πρέπει να περάσει στου ανθρώπου. Αυτό σημαίνει η κοινωνική οικονομία τη αγορά. Και γι' αυτό μιλάμε για τον κοινωνικό πυλώνα, ένα πυλώνα ο οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλα αυτά σημαίνουν στεναρότερη υποστήριξη και σημαίνουν ότι είναι σωστό να εργαστούμε για όλα αυτά τα θέματα με φιλοδοξίε, με στοχοπροσύλωση. Βεβαίω και δεν θα είμαστε ποτέ τέλεια, αλλά η προσπάθεια να βελτιωθούμε, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένα θέματα στον κοινωνικό πυλώνα, αυτή η προσπάθεια πρέπει να είναι ο ε, ανώτερος και ανώτατος στόχο μα. Οι στόχοι τη βιωσιμότητα. για μα είναι κατευθυντήρια γραμμή. Η βιωσιμότητα και οι στόχοι τη βιωσιμότητα είναι προ το συμφέρον όλων μα. γιατί εντωμεταξύ όλοι κατανοήσαμε ότι ότι το ρολόι χτυπά, ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος, ότι ο πλανήτης μας χρειάζεται βοήθεια, ότι αυτός ο κόσμος που ζούμε είναι η βάση της περαιτέρω επιβίωσης. Και όλα αυτά πρέπει να γίνουν μέσα σε ένα καλό, φιλικό, περιβάλλον, απέναντι στο κλίμα. Ως εκ τούτου λοιπόν οι στόχοι της ε, βιωσιμότητας ε, εξυπηρετούν όλους μας και γι' αυτό οφείλουμε να τους επιδιώξουμε με όλη τη δύναμή μας. Όσον αφορά ε, τις δύο φάσεις ε, και τα δύο βήματα ε, πρέπει να ακολουθήσουν παράλληλα. Γιατί αυτά που είπα σημαίνουν ότι πράγματι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές. Γνωρίζουμε όμως ότι παράλληλα μπορούμε να επιφέρουμε και αλλαγές ε, σε αυτό τον πλανήτη των μεγάλων παικτών. Εκεί η Ευρώπη μπορεί να καταλάβει μια θέση και πρέπει να την καταλάβει για να προωθήσει τις αλλαγές. Στη συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα για πρώτη φορά ενώθηκαν όλες οι δυνάμεις. Γι' αυτό λοιπόν ας επανέλθουμε σε αυτές τις δυνάμεις με αυτό το πνεύμα να προχωρήσουμε για να αντιμετωπίσουμε ένα από τα πιο επίγοντα προβλήματα που μας έχουν, που μας έχουν πλήξει. Άλλο επίγον θέμα, το θέμα της ψηφιοποίησης. Και εκεί χρειαζόμαστε ενωμένες δυνάμεις. Και εκεί χρειαζόμαστε αφενός τις δυνάμεις που πρέπει να είναι σε θέση την ψηφιοποίηση, να την αντιμετωπίσουν με ενθουσιασμό, να ενισχύσουν την οικονομία, να προσφέρουν πολλές δυνατότητες. Από την άλλη όμως να διατηρηθεί και η κοινωνική οικονομία της αγοράς μέσα σε ένα ηθικό πλαίσιο. Το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, ε, το θέμα της συμπεριφοράς στον κυβερνοχώρο. Αυτά τα δύο θέματα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με σύνεση, με μέτρο και στην ε, κυβερνοασφάλεια και ως Ευρώπη πρέπει να προχωρήσουμε, να γίνουμε πιο ισχυροί. Γιατί στην κυβερνοασφάλεια ελοχεύουν πολλοί κίνδυνοι που μπορούμε να τι αντιμετωπίσουμε μόνο αν είμαστε ενωμένοι. Υπάρχουν κίνδυνοι που είναι σημαντικοί για την οικονομία αλλά και για την κοινωνία. Και κανένα κράτο δεν είναι σε θέση μόνο του να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Μόνο από κοινού μπορούμε να επιφέρουμε ασφάλεια στην Ευρώπη που αξίζει στην Ευρώπη. Ο άνθρωπο μέσα στην ψηφιοποίηση. Αυτό είναι το πιο ευγενέ καθήκον τη κοινωνική οικονομία τη αγορά. Να μπορεί κανεί να εργάζεται, αλλά παράλληλα να απολάβει και προστασία, ε, Αυτό βέβαια εξαρτάται από τις συνθήκες εργασίας που πρέπει τώρα να μάθουμε όλα αυτά να τα μεταφέρουμε σε ένα ψηφιακό κόσμο. Ο click worker, ο cloud worker, ο άνθρωπος που εργάζεται σε πλατφόρμες ε, και σε αυτόν θα πρέπει να ισχύουν όλες οι προστασίες που πρέπει να επιφέρουμε από κοινού. Γι' αυτό λοιπόν κυρίες και κύριοι πρέπει να σας πω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ενδιαφέρον σας άκουσα. Κύριε Μόιτεν, ακούγοντας εσά, ε, πρέπει να σα πω, ανακουφίστηκα. Ανακουφίστηκα που δεν θα με ψηφίσετε. Για μένα αυτό είναι ό,τι καλύτερο είχα να ακούσω σήμερα το πρωί. Υπάρχει κάποιο αίτημα για παρέμβαση κατά την έννοια ε, από τον κύριο Σένσροτ. Θα ήθελα να αναφερθώ στο παράτημα 7, άρθρο 1, όπου γίνεται λόγο για τη δημοσιοποίηση των οικονομικών συμφερόντων και άρθρο 2, καλό το Κοινοβούλιο να εξετάσει κατά πόσον υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Και έχω ήδη μία πρόταση το τι μπορεί και πρέπει να γίνει. Α, έτσι να γίνει. Όπως με βλέπετε εμένα. Στρέψτε το βλέμμα προς εμένα και δέστε το τι ακριβώς εννοώ. Ε, ε, ε, πρόεδρος, κοιτάξτε σας παρακαλώ πάρα πολύ να καθίσετε. Θα συνεχίσουμε γιατί αυτό δεν είναι πραγματικό διαδικαστικό. Κύριε Γκάσπαρη, έχετε το λόγο. Για δύο λεπτά, κύριε Γκάσπαρη. Αξιότιμε Πρόεδρε, εμείς ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και ως Ευρωπαίοι Χριστιανοδημοκράτες μπήκαμε στην προεκλογική εκστρατεία με τον κύριο Βάμπα και Βίμπα και θέλουμε και θέλαμε μάλλον να γίνει πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όμως το Συμβούλιο, ορισμένοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ποδοπάτησαν τη βούληση των πολιτών. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπήρξαν πολιτικές ομάδες που δεν είχαν το θάρρος όπως έγινε πριν από πέντε ε, χρόνια να στηρίξουν τον Spitzenkandidat που είχαμε προτείνει. Κυρία Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σα έχουμε σήμερα εδώ στην Ολομέλεια και μέχρι τι 6 ώρα το απόγευμα θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εκλεγείτε πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουμε δύσκολε καταστάσει και εσεί έχετε μπροστά σα ένα τεράστιο πακέτο καθηκόντων. Τα τελευταία χρόνια, οποτεδήποτε είχαμε δυσκολίε, εμεί εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήμασταν σε θέση διακομματικά, ε, όχι βέβαια με όλε τι πολιτικέ ομάδε, γιατί δυστυχώ υπάρχουν και λαϊκιστέ και ακραίοι που δεν θέλουν να εξελιχθεί περαιτέρω η Ευρώπη, αλλά θέλουν να την καταστρέψουν. Εν πάση περιπτώσει, διακομματικά κατορθώσαμε να ε, καταλήξουμε σε συμβιβασμού για να στηρίξουμε αυτή την Ήπειρο και να την εξελίξουμε περαιτέρω προ όφελο των πολιτών. Σα παρακαλώ να απευθυνθείτε σε αυτό το κοινοβούλιο που είναι πάνω από το ίμιση των πολιτών που ψήφισαν. Αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να το θεωρείτε ότι είναι εταίρο οποτεδήποτε θέλετε να προχωρήσετε στην Ευρώπη οποτεδήποτε θέλετε να σπάσετε αποκλεισμού στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εμεί πάντα ήμασταν η αιχμή του δόρατο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλω να πιστεύω ότι και εσεί θα παραμείνετε μαζί με εμά στην αυτή την αιχμή του δόρατο. Κύριε Μόιτεν, αυτά που είπατε σήμερα προσβλητικά, ε, γεμάτα μίσο, ε, ε, συκοφαντήσατε την κυρία Φοντελάν. Χτε το βράδυ δεν μπορέσατε ούτε καν να γίνετε πρόεδρος στη δική σας την περιφέρεια. Εντάξει, καταλαβαίνουμε την απογοητευσία σας, αλλά τι φταίει η κυρία Φαντελάνη. Η κυρία Φαντελάνη δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Αλλού να χύσετε το δηλητήριό σας. Ευχαριστώ πολύ. Δύο λεπτά ο κύριος Γκουαλτιέρη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Φοντερ ο ορισμός σας ε, είναι αποτέλεσμα ε, μιας ε, δύσκολης εμπλοκής στην, στο Συμβούλιο που δεν κατάφερε να προωθήσει την θέση του Spitzenkandidat. Πρόκειται για μια διαδικασία που προβλέπεται από τους κανονισμούς αλλά θεσμικά αποτελεί πλήγμα, αποτελεί μια πληγή την οποία θα πρέπει να κλείσουμε έτσι ώστε να μην δημιουργήσει πρόβλημα στην οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή δημοκρατίας. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό η ομάδα μας, όπως και άλλε ομάδες, ε, είναι σημαντικό, λέω, που να ξεκινήσει μία ε, πραγματική πολιτική ε, συζήτηση. Πρόκειται για κάτι που ξεκινήσαμε εδώ και που μπορεί να ενισχύσει την σχέση με τους Ευρωπαίους πολίτες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από όλους, κυρίως δε από το Συμβούλιο. Στην επιστολή σας, στην ομάδα μας και στα ωραία λόγια που είπατε. Εσείς απαντήσατε θετικά σε πολλά από τα αιτήματά μας για πιο σοβαρούς ε, και φιλόδοξους στόχους, ε, για περισσότερες δημόσιες επενδύσεις και το τονίζω αυτό καλή χρήση της ευελιξίας έτσι ώστε να υπάρξει υποστήριξη της ανάπτυξης, ε, ε, ελάχιστη ε, αμοιβή, εγγύηση για τους νέους, κοινή φορολόγηση για τις επιχειρήσεις, ανθρωπιστικούς διαδρόμους, συμμαχία και για το περιβάλλον, καθώς επίσης και μία σειρά από σημαντικά θέματα μεταξύ θεσμικά μεταξύ των οποίων και η ενίσχυση του θεσμού του Candidate. Εμείς θα αγωνιστούμε ε, με πεποίθηση για την υλοποίηση των στόχων αυτών. Από την επιστολή σας και από τη συζήτηση εδώ μου φαίνεται ότι ε, καταλήγουμε ότι οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις είναι αυτές οι οποίες, με τις οποίες θα συζητήσετε και όταν θα είστε ενδεχομένως στην Επιτροπή. Ε, μόνο με τις φιλοευρωπαϊκές και χωρίς κανέναν άλλον. Οι λαϊκιστές και οι εθνικιστές έχουν θέσεις οι οποίες δεν μας αφορούν. Κυρία Φόντερ Λάγεν, ε, θα είναι η πολιτική μας ομάδα προσεκτική, ε, προσεκτικός και απαιτητικός συνομιλητής. Εμείς ε, δεν αρκούμαστε στα λόγια. Εάν αν μετά τα λόγια δεν ακολουθήσουν πράξεις, δεν θα έχετε την υποστήριξή, σας, υποστήριξή μας. Εάν αντιθέτως ε, συγκεκριμενοποιήσετε αυτά τα οποία μας είπατε, μπορείτε να βασίζεστε ε, στην ε, επαγρύπνησή μας, αλλά στην συμμετοχή μας σε αυτή τη διαδικασία για μια καλύτερη και δικαιότερη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζουρνέ, ένα λεπτό. Είναι πολύ λίγο ένα λεπτό. Εμείς θα πούμε ότι θα σας υποστηρίξουμε έτσι ώστε να ε, έχετε σε αυτό το φύλλο ευρωπαϊκό ημικύκλιο μια ε, ικανοποιητική πλειοψηφία. Ε, είχαμε, πήγαμε σε εκλογές στις οποίες οι λαϊκιστές, οι εθνικιστές έλεγαν ότι σίγουρα θα έχουν την πλειοψηφία. Δεν έγινε αυτό. Οι προτάσεις σας είναι πολύ σωστές. Τις διαβάσαμε όλοι. Ε, και στις ε, προτάσεις σας ε, βρήκαμε και κάποιες από τις δικές μας θέσεις για το κλίμα, η ουδετερότητα, η κλιματική, ο φόρος για το διοξίδιο του άνθρακος, για τις εκπομπές, οι κοινωνικές αρχές οι οποίες μας βρίσκουν σύμφωνους. και νομίζω ότι βρίσκουν σύμφωνους και όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτήν την φιλοευρωπαϊκή διαδικασία. Ε, βεβαίως, οι, οι, οι εμπορικές συμφωνίες ε, είναι σημαντικές, με ρήτρε συγκεκριμένες, ε, η δέσμευση για την υλοποίηση των αρχών των Παρισίων. Σε αυτό το ημικύκλιο χρειαζόμαστε το σύνολο των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων γιατί είναι πολλοί αυτοί που μας λένε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα του κλίματος, είναι επίγουσα η διαδικασία, ναι, συμφωνούμε, συμφωνούμε, αλλά εδώ σήμερα στο ημικύκλιο αυτοί που ε, συνεχώς κηρύττουν ε, την επίγουσα ε, κλιματική διαδικασία ενώ βλέπουν συγκεκριμένες προτάσεις δεν ενστερνίζονται τις προτάσεις αυτές, δεν αναλαμβάνουν κάποια δέσμευση. Καλό λοιπόν όλους να δείξουν υπεύθυνη θέση. Καλό όλους να δεσμευτούν γύρω από εσά και γύρω από μια φιλοευρωπαϊκή πλειοψηφία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκίγκολτ, 1,5 λεπτό παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ Φοντερ Λάιν, μας ε, προσφέρατε ε, μια πράσινη συμφωνία, ένα Green Deal, ε, καλός ο τίτλος, αλλά δεν έχει αρκετό πράσινο περιεχόμενο. Ο κόσμος αντιμετωπίζει δύο μεγάλες οικολογικές κρίσεις. Την ε, κρίση του κλίματος ε, και την εξαφάνιση των ειδών. Όσον αφορά την κρίση του κλίματος, είπαμε στο Κοινοβούλιο, μέχρι το 2030 πρέπει να έχουμε ένα μείον 55%. Εσείς σήμερα δεν είπατε ότι οθετείτε αυτό το στόχο, αλλά αυτό είναι το μέτρο. Αυτό είναι το κριτήριο που ζητούν να εφαρμόζεται το ζητούν οι νέοι, το ζητά και η επιστήμη. Χρειαζόμαστε λοιπόν μία σαφή δέσμευση μείων κατά 55% εκπομπές ε, θερμοκηπίων, εκπομπές θερμοκηπίου μέχρι το 2030. Και το δεύτερο είναι η εξαφάνιση των ειδών. Ε, ζήσατε μεγάλο χρονικό διάστημα στο Ανόβερο. Εγώ εκεί παλαιότερα μέτραγα τις ε, πεταλούδες και πολλά άλλα ζώα που σήμερα όμως πια δεν υπάρχουν. Δεν είπατε τίποτα για την κρίση της βιοπικιλότητας. Εμείς λοιπόν ζητάμε με σαφήνεια μια νέα αγροτική πολιτική που θα προστατεύει τους γεωργούς ε, και θα παρεμποδίζει την εξαφάνιση ειδών. Σήμερα να δεσμευτείτε ότι θα εφαρμόσετε μια τέτοια γεωργική πολιτική που θα προστατεύει το κλίμα και επιτέλους ε, θα βάλει τέλος ε, σε αυτή την ταχύτατη εξαφάνιση ειδών. Και να πω και κάτι άλλο. Στα ευρωπαϊκά εξωτερικά σύνορα δεν κατέστη δυνατόν να αποφύγουμε τελείως του τους θανάτους. Και σας ερωτώ, είσαστε ε, πρόθυμοι να ε, θεσπίσετε ευρωπαϊκή ακτοφυλακή. Η ομιλία σας ήταν καλή, αλλά το περιεχόμενο που θίξατε δεν ήταν ικανοποιητικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ να σέβεστε τον χρόνο αγόρευσης, γιατί είναι πάρα πολλοί οι ομιλητές. Ο κύριος Τζάνι, δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ε, κύριε Υπουργέ Βόντερ Λάιν. Η εισήγησή σας δεν μας ε, εξέπληξε. Είναι λόγια τα οποία έχουμε ακούσει πολλές φορές εδώ σε τούτο το ημικύκλιο ε, με πλήθος ε, υποσχέσεων που ξέρετε ότι δεν θα μπορέσετε να τηρήσετε. Την πορεία την είδαμε τις τελευταίες μέρες αλλά και στην Ολομέλεια. Δηλαδή πρέπει να ισορροπήσετε δύο διαφορετικά στοιχεία, δύο διαφορετικές πλευρές, διαφορετικά συμφέροντα από τη μία με την δεξιά με μια πιο ορθολογική προσέγγιση και για τη μετανάστευση ε, και για την ε, οικονομία αλλά από την άλλη την αριστερή που έχει ιδεολογική προσέγγιση υποδοχής ε, χωρίς διάκριση και μια πολύ φανατική προσέγγιση όσον αφορά το κλίμα. Θα πρέπει λοιπόν η κεντροδεξιά να αποφασίσει εάν ε, ε, θέλει να υποχωρήσει απέναντι στις απειλές ε, της αριστεράς, έτσι φάνηκε να θέλετε να κάνετε εσείς, ή θα προτιμήσετε μία λογική, ορθολογική προσέγγιση η οποία θα δώσει την δυνατότητα στην Ευρώπη να βγει από την κρίση. Μια κρίση στην οποία την έβαλαν οι κακές πολιτικές. Εσείς μιλήσατε για υποδοχή, μιλήσατε για διάσωση στη θάλασσα Πολύ όμορφα είναι όλα αυτά τα λόγια. Ωστόσο, θα πρέπει να τα πείτε αυτά στους ε, χιλιάδες, ε, στα εκατομμύρια των Ευρωπαίων που υποφέρουν από τις, ε, τα αποτελέσματα των πολιτικών που έχουν κάνει αυτές οι πολιτικές ομάδες. Όταν θα πρέπει να τα πείτε σε αυτούς που έχουν υποφέρει από τις καταστροφικές πολιτικές. Ε, θα πρέπει να δείτε εάν έχετε μία πλειοψηφία η οποία ε, θα μπορέσει να προχωρήσει σε αυτήν την τόσο ριζική, ριζοσπαστική αλλαγή που ζητούν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Δεν είναι δυνατόν να λέτε ότι αυτοί που έχουν διαφορετική άποψη δεν θα βοηθήσουν εσάς να κυβερνήσετε, δεν θα βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να προχωρήσει, δεν θα βοηθήσουν έτσι ώστε τα επόμενα χρόνια να έχουμε ανωδική πορεία. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι αντιπροσωπεύετε ή μπορείτε να αντιπροσωπεύσετε την πρόοδο που χρειαζόμαστε, την αλλαγή που χρειαζόμαστε. Δεν είναι δυνατόν να υποστηρίξουμε μία πολιτική συμμαχία η οποία στην ουσία μπάζει από παντού. Μία πολιτική που είναι σουρωτήρη. Ε, νομίζω ότι κανένας ε, δεν έχει ε, εδώ πραγματικά και με την καρδιά για του ε, δώσει το πράσινο φως για αυτήν την προεδρία. Ε, απλώς λογικά σκεπτόμενοι οι μεν λένε ότι θα πρέπει να κάνουμε την καρδιά μας πέτρα και να προχωρήσουμε έτσι και οι άλλοι το αντίθετο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Φοντελάγκ. Στην πολιτική αντιλαμβανόμαστε ότι πολλέ φορέ πρέπει να δημιουργηθεί η πλειοψηφία. Αλλά είναι σημαντικό τι υποσχέσει κάνετε και μέχρι πού φτάνετε με τι υποσχέσει. Ω ένα σεφ σε ένα μεγάλο εστιατόριο, είστε υπεύθυνοι για τα συστατικά που θα βάλετε στο φαγητό και ποια θα είναι η γεύση του φαγητού και πώ θα του αρέσει στου πελάτε. Και σε πέντε χρόνια, νομίζω, οι πολίτε στη Ρήγα και σε μικρά χωριά της Πορτογαλίας θα πρέπει να πούν ε, αυτό ήταν καλό αποτέλεσμα. Δεν νομίζω να ισχύει όμω αυτό. Γιατί? για την περασμένη εβδομάδα ήρθατε στην ομάδα μα και είπατε ότι μία από τι αρχέ ήταν η επικουρικότητα. Σήμερα υπολόγισα, είναι η πρώτη φορά που το είπατε στα 30 λεπτά. Δεν ξέρω ότι η διακρατική ω κατάλογο ε, θα είναι στην καρδιά των πολιτών. Δεν νομίζω ότι αυτό θα είναι καλό για όλου. Και ποια είναι τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Ε, λοιπά Λυπάμαι. Είναι μια απογοήτευση ε, σήμερα σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα αυτά που άκουσα. Ο κύριος Φερέιρα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Βαντερνάιεν. Εσείς ε, προσπαθείτε να μας πείτε όμως ότι υπάρχουν προβλήματα ανασφάλειας εκατομμυρίων χιλιάδων εργαζομένων. Ε, υπάρχουν και ανισορροπίες ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες στο χώρο της εργασίας. Το πρόβλημα του κεφαλαίου, το πρόβλημα των κοινωνικών δικαιωμάτων, όλα αυτά πλήττονται. Ε, το πρόβλημα των πολυεθνικών, ε, των πολέμων, η Ευρώπη της πρόοδου, από την άλλη πλευρά της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ε, πράσπισης του κλίματος, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, της ειρήνης. Όλα αυτά είναι αξίες που τις ε, στηρίζεται, αλλά δεν μπορούν να ε, ξεκινήσουν από την συνένεση που έχουμε μπροστά μας. Γι' αυτό θα πρέπει να κάνετε μια επιλογή. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ε, δουλέψουμε για αυτό το μέρος της Ευρώπης και της επόμενης. Και εσείς θα πρέπει να κάνετε αυτή τη συμφιλίωση ανάμεσα σε αυτές τις δύο ε, αξίες. Κύριο Σόνεμπορν. Ενάμιση λεπτό ο κύριος Σόνεμπορν. Αγαπητή ε, κυρία Φόντερ Λάιεν, καλώς ορίσατε. Χαίρομαι που δεν είμαι πλέον ο μόνος ε, που δεν εκπροσωπώ τη μη σοβαρή δημοκρατία. Ε, το ότι θα επανέλθει ο κύριος Μπορέλ ε, γιατί είχε ξεχάσει να αναφέρει τις 300.000 ευρώ καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι σωστό. Δεν μπορεί να εκπροσωπεί το κόσμο. Η Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία επίσης έχει καταδικαστεί για πιστία δημόσιου χρήματος ε, και ακόμα δεν έχει υπάρξει ποτέ ε, κεντρικός ε, τραπεζίτης. Υποτίθεται θα είναι πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ένας Βέλγος που ούτε στο Βέλγιο δεν μπόρεσε να σχηματίσει κυβέρνηση και να γίνει πρόεδρος του Συμβουλίου. Ένας άνθρωπος ο οποίος προσπάθησε να συμβάσει καταστάσεις και επιπρόσθετα και εσείς κυρία Φόντερ η οποία δεν έχετε ιδέα για ευρωπαϊκά θέματα. Απλά ήσασταν υπουργό και κατηγορήστε για ε, κακοδιαχείριση, ε, για διάτρητα οικονομικά. Υπάρχουν λοιπόν ε, αυτές οι υποψηφιότητες και γι' αυτό το λόγο εσείς έρχεστε σε επαφή με τον Όρμπαν, τον Σαλβίνη δεν πρέπει λοιπόν να αφήσουμε την Ευρώπη στους αδαείς. Αυτά είχα να πω. Κύριε Ντότς, για δύο λεπτά. Αγαπητή κυρία Φόντερ Λάιεν, θα ήθελα να σας πω τα εξής εκ μέρους του ΕΛΚΑ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει τα πάντα για να προστατεύσει τα ευρωπαϊκά σύνορα. Πρέπει να σταματήσει η μετανάστευση και μπορεί να σταματήσει μόνο εάν δεν δεχόμεθα τους παράτυπους μετανάστες οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά μας και τον παραδοσιακό τρόπο ζωής. Η νέα πρόεδρος Επιτροπής ε, κατ' εμάς οφείλει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και να εκτιμήσει τις προσπάθειες που κάνουν αρκετά κράτη για να προστατεύσουν τα εξωτερικά σύνορα. Ε, το άρθρο 2 στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει το εξής ε, ισότητα των κρατών μελών και διαφύλαξη της ε, εθνικής ταυτότητας γιατί αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο. Τα τελευταία χρόνια η αριστερή πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η πλειοψηφία λοιπόν αυτή ε, χρησιμοποιώντας ε, το άρθρο 7 ε, θέλησε να άρει κάποια παγιωμένα δικαιώματα. Εμείς λοιπόν περιμένουμε από τη νέα πρόεδρο της Επιτροπής όπως σας είπα, να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να διαφυλάξει την εθνική ταυτότητα και την ε, συνταγματικά νόμιμη συμμετοχή των ε, κρατών μελών. Όταν πρόκειται για, τις ε, περιφερειακές, όταν πρόκειται για την περιφερειακή ανάπτυξη, αυτά που δίδονται στις περιφέρειες και στις χώρες δεν είναι δωρεά δεν είναι χάρη. Πρόκειται για ένα βασικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατ' ουσίαν πρόκειται για την περιφερειακή σύγκληση και για το λόγο αυτό οι επενδύσεις είναι απαραίτητε σε ορισμένες χώρες. Περιμένουμε λοιπόν από τη νέα πρόεδρο, περιμένουμε ο νέος προϋπολογισμός να μην τιμωρεί τις χώρες εκείνες που αυτή τη στιγμή είναι φτωχότερες. Οφείλουμε να διεκδικήσουμε την μεγαλύτερη σύγκληση, γιατί ε, οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης είναι εκείνες κυρίως που υποφέρουν. Η κυρία Ντάλη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα επόμενα πέντε χρόνια θέλουμε ηγεσία. Αυτό όμως δεν είναι υπεπατημένη από το σημείο της αφετηρίας. Θέλουμε μια ε, κομισιόν που να είναι φιλόδοξη, προοδευτική και να μην αντιστέκεται στις αλλαγέ. Είναι θετικό το οποίο θέλετε να κάνετε ουδέτερη την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2050 και ότι έχετε δεσμευτεί να γίνει αυτό νόμος τις πρώτες 100 σας μέρες. Αλλά όταν πρόκειται για τον στόχο το 2030 να έχετε κατά νου ότι αυτό το σώμα ζήτησε για αυτό το στόχο του 55% γιατί αυτό ε, συνάδει με τη μακροχρόνια στρατηγική και με τους στόχους του Παρισίου. Μιλήσατε για την παράταση του ETS. Ε, η αεροπορία και οι θαλάσσιες μεταφορές πρέπει να συνεισφέρουν, αλλά το ETS δεν μπορεί να ε, επεκταθεί στις μεταφορές γενικά δουλέψαν πολύ σκληρά για αυτού του στόχου. Γι' αυτό ζητήσαμε για μια σαφή δέσμευση ότι δεν θα επαναχωρήσετε από το πρότυπα του και το, το, τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα. Θέλουμε να δεσμευτείτε για μια στρατηγική βιοπικιλότητα και θέλουμε να κατανοήσουμε τη θέση σα για την στατική για το μη τοξικό περιβάλλον. Ε, θέλουμε μια ανανέωση της βιομηχανικής πολιτικής. Να μην εστιάζεται μόνο στη ψηφιοποίηση και την αυτοματοποίηση, αλλά να περιλαμβάνει και την οικολογική πτυχή. Μια βιομηχανική πολιτική που να λαμβάνει υπόψη τους εργαζόμενους, τους μελλοντικούς εργαζόμενους, τους φοιτητέ και τους νέους μας. Και επιτρέψτε μου να πω και κάποια λόγια για τη μετανάστευση. Μιλήσατε για μια νέα κίνηση στο θέμα της μετανάστευσης. Ως ε, μέλος ε, ε, του Ευρωκοινοβουλίου από τη Μάλτα θέλω να θέσουμε την μετανάστευση ως προτεραιότητα όπου η αλληλεγγύη να μην είναι απλά ένα σύνθημα αλλά όπου οι νομοθετικές προτάσεις όπως ο κανονισμός του Δουβλίνου να θεσπιστούν και να γίνουν νόμοι έτσι ώστε όχι μόνο μερικές πόλεις και χώρες να επομίζονται το βάρος όπως γίνεται σήμερα. Θέλουμε πολιτικές που να αλλάζουν τα πράγματα αν θέλουμε να προχωρήσουμε και αυτές είναι οι πολιτικές που εμείς ως σοσιαλιστές και δημοκράτες θα προωθήσουμε. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, η κυρία Βόουτεν τώρα. Ευχαριστώ μαζί με άλλου προλαλήσαντε τη Renew σκέφτηκα ε, θα στήριζα την κυρία Φόντελάιν σήμερα. Το σύστημα που την έχει θέσει ενώπιον μα είναι ε, διασπασμένο. Αλλά μπήκα ε, σε αυτό το σώμα από εκατομμύρια Βρετανού που πιστεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ζητούν τα καλύτερα από την Ευρώπη και που μα θέλουν να παραμείνουμε εδώ. Εμείς θα ήμασταν ανόητοι να χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Χρειαζόμαστε δράση και όχι μία αναποφασιστικότητα. Κύριε σα λέω ότι η ψήφο μα δεν έρχεται εύκολα. Αν θα σα στηρίξω είναι ένα τίμημα που ζητάω εγώ από τη στήριξή σα. Θα έπρεπε να αναμορφώσετε αυτό το σύστημα. Θα πρέπει να δεσμευτείτε για πραγματική δράση και όχι μόνο λόγια για την, το θέμα του κλίματος. Θα έπρεπε να αρχίσετε άμεσα τη μεταρρύθμιση τη διαδικασία του Δουβλίνου. Και για μένα το θέμα είναι να χρησιμοποιήσετε την επιρροή σα σε κάθε τράπεζα διαπραγματεύσεων έτσι ώστε να ζητήσετε μια μακρά παράταση έτσι ώστε η Βρετανία να παραμείνει παραμείνει μέρος αυτής της ευρωπαϊκής οικογένειας. Ο κύριος Eichhout, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Βαντερ Λάγεν, ευχαριστώ για το όσο μας είπατε. Σε ε, σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα έχετε κάνει ένα τεράστιο βήμα. Αλλά αναρωτιόμαστε για ποιον θα ψηφίσουμε. Υπάρχουν τόσο μεγάλες αλλαγές ε, ε, και τόσο μεγάλη ασάφεια. Θα είναι μείον 50, μείον 55 όσον αφορά το κλίμα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να βάλετε και κάποια συγκεκριμένη εκκίνηση Δεκέμβριο του 20. Ακόμα αυτό είναι ασαφές. Ε, επίσης για τη γεωργική πολιτική, τι θα κάνετε με την παρούσα μεταρρύθμιση των γεωργικών πολιτικών. Ε, επίσης, τι ε, σημαίνει το ETS και η, μετα... η μεταρρύθμιση του. Αυτό Έχω την εντύπωση ότι εδώ παίζεται λίγο το παιχνίδι της γερμανικής αυτοβιομηχανίας, αυτοκινητοβιομηχανίας. Τέλος, ε, για το κράτος δικαίου, πολύ ωραία τα λόγια, αλλά συγκεκριμένη δράση. Εσείς θα υποστηρίξετε το Κοινοβούλιο στη διαδικασία του άρθρου 7 κατά της Ουγγαρίας. Συγκεκριμένα πράγματα. Ναι ή όχι. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Μπέ για ένα λεπτό. Κυρία Βόντερ Λάγεν, ε, ε, σε αυτό το ημικύκλιο στο οποίο θέλετε, ε, ε, ε, εδώ στο Κοινοβούλιο ο κύριος Γιούνκερ, τον οποίον θέλετε να διαδεχθείτε, είπε ότι είμαστε στην τελευταία ευκαιρία που είχαμε. Χρειάζεται ευρωπαϊκή, λέει, συνεργασία. Αλλά τελικά στην πλάτη των λαών προχώρησαν οι διορισμοί των, στις υψηλές θέσεις των οργάνων και βρίσκεστε εσείς εδώ σήμερα γιατί κάποιες πολιτικές ομάδες σας έσπρωξαν ε, και μιλάμε για το παγκοσμιοποιημένο εμπόριο, το μιλάτε εσείς για το παγκοσμιοποιημένο εμπόριο το οποίο καταστρέφει τις οικογένειές μας και τις θέσεις εργασίας μας. Ε, σπρώχνεται ακόμα παραπέρα το θέμα όσον αφορά αυτή την ε, παράλληλη θέση όσον αφορά την χαλαρή συγγνώμη θέση όσον αφορά το μεταναστευτικό και λέτε να πάμε ακόμα πιο πέρα. Θέλετε να παίξετε το παιχνίδι της αριστεράς ε, και για όλους αυτούς τους λόγους, για να πάρετε εσείς τους ψήφου της αριστεράς, δεν θα έχετε τις δικές μα ψήφου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Λούντκριν. Κυρία Φαντελάιεν. Πιστεύετε για την, τις Ηνωμένε Πολιτείε της Ευρώπης, αλλά αυτό είναι σε αντίθεση με τον επιθυμούν οι πολίτες ε, να καθορίσουν μόνοι τους ε, το μέλλον τους. Γιατί αν συμβεί κάτι τέτοιο, πάρα πολλοί θα χάσουν πάρα πολλά δικαιώματα και η κοινή λογική απαιτεί τα κράτη-μέλη στην Ευρώπη να συνεργάζονται μεταξύ τους, να μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις. Μία κεντρική πολιτική ένωση ε, δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει ισοπαίδωση, γιατί πολίτες και τα κράτη θέλουν να διαφυλάξουν την ε, ιστορία τους ε, και τον πολιτισμό τους. Αυτό που πρέπει να υποστηρίξουμε είναι κάθε πολίτης να μπορεί να έχει τις δικές του τις φιλοδοξίες ακούγοντας την ομιλία σας σήμερα το πρωί ε, κατάλαβα απόλυτα ότι δεν είσαστε κατάλληλοι για τη δουλειά του Πρόεδρου της Επιτροπής και γι' αυτό θα σας ε, καταψηφίσουμε. Ένα λεπτό, Ματίας. Κυρία Πάντα Λάιν, φαντάζομαι ότι θα έχετε καταλάβει ότι υπάρχουν πολιτικές ομάδες οι οποίες δεν συμφωνούν με την υποψηφιότητά σας. Υπήρξαν και υποψηφιότητες ε, οι οποίες αποκλείστηκαν όσον αφορά το αξίωμα του Πρόεδρου της Επιτροπής. Πρέπει να γίνουν κάποιες επιλογές και γι' αυτό ερωτώ. Υπάρχουν χώρες ε, οι οποίες ε, έχουν πλεόνασμα. Τι θα γίνει με, τις, με το πλώνισμα αυτό. Είτε θα επενδύσουμε στον πλανήτη, είτε θα επενδύσουμε στη στρατιωτικοποίηση. Εσείς υπέρ ποιας επιλογής θα ταχθείτε ή όσον αφορά τις offshore θα τις αντιμετωπίσουμε. Εσείς υπέρ οποίου πράγματος θα ταχτείτε υπέρ των δικαιωμάτων των εργαζομένων ή θα συνεχίσετε να ε, καταστρέφετε τα δικαιώματα αυτά. Ε, θα έχουμε μία πολιτική υποδοχή των μεταναστών. Εσείς από ποια πλευρά είστε, κυρία Φοντερ Λάιν. Ε, χρειαζόμαστε σαφείς επιλογές δεν νομίζω ότι ήταν καλό το ότι υπήρξαν αυτές οι δύο εβδομάδες αντιφατικών συζητήσεων. Γιατί αν εκλεγείτε τελικά φοβάμαι ότι θα υπάρξει άλλη μία απογοήτευση. Κυρία Μπεγκίν. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, ε, κοιτάξτε, εγώ ε, ω μητέρα τριών παιδιών χαίρομαι πάρα πολύ που για πρώτη φορά βλέπω μια γυναίκα η οποία προτείνεται να προεδρεύσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό χωρίς αμφιβολία είναι κάτι το ευχάριστο, αλλά δεν θέλω αυτή να είναι και η μόνη αλλαγή, γιατί οι κυβερνήσεις που στήριξαν την υποψηφιότητά σα ε, προφανώ είδαν σε εσά έναν καλό πρόεδρο, αλλά ήθελαν ε, κυρίω να πούν όχι σε αυτού που είχαν την έπαρση να πιστεύουν ότι θα γινόντουσαν απολύτω αποδεκτέ οι υποψηφιότητε αυτέ. Εγώ θέλω να πω ότι σε αυτή την Ευρώπη, αν θέλουμε να ζούμε μαζί, θα πρέπει να αποφασίζουμε μαζί, όλοι μαζί. Κυρία Φοντελάν, μετά τη συνάντησή μα, ε, υιοθετήσατε τα στοιχεία του προγράμματός μας για τον κατώτατο μισθό, μια νέα συμφωνία για τη μετανάστευση, φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις για το κλίμα και επιτέλους να υπάρχουν εγγυήσεις για την νομοθετική πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό ε, οι πέντε αστέρες θα σας στηρίξουν, αλλά κατά τα επόμενα πέντε έτη θα πρέπει να αποδεικνύετε ότι αξίζεται αυτήν την εμπιστοσύνη μας. Εμείς θα συνεχίσουμε να σας ελέγχουμε και να ε, ερχόμαστε σε σκληρή αντιπαράθεση αν δεν προασπίζεστε τα συμφερόντα των Ευρωπαίων πολιτών. Ε, δεν χρειάζεται να είναι κανείς ε, Γάλλος, Ευρωπαίος, Γάλλος, Γερμανός, Ιταλός, Ισπανός για να έχουμε μια καλή Ευρώπη. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να δείξουμε στον κόσμο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι απλά το άθροισμα των κρατών. Κυρία Φοντελάιν, αν θέλετε να υπάρξει μια πραγματική αλλαγή, να επιφέρει την αλλαγή που αξίζει στους Ευρωπαίους πολίτες να μην τους απογοητεύσετε. Ο κύριος Γκονζάλες Πόνς. Δύο λεπτά. Όλοι ε, διαπίστωσαν ότι δεν ήταν σωστός ο τρόπος με τον οποίο το Συμβούλιο αντιμετώπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και ο τρόπος με τον οποίο σας όρισε εσάς. Αλλά αναγνωρίζουν όλοι ότι είναι η χειρότερη στιγμή ε, για να υπάρξει θεσμική κρίση. Δεν είναι δυνατόν να παίξουμε το παιχνίδι των ακραίων και λαϊκιστών. Το Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να κάνει λάθος. Γι' αυτό εμείς θα σας εμπιστεύουμε εμπιστευτούμε. Ε, έχουμε ε, μια Ευρώπη η οποία δεν μπορεί να είναι ακέφαλη ε, μέσα σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει τόσα προβλήματα εμπορικά, κοινωνικά και άλλα. Εσείς είστε δεσμευμένοι στην οδό της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Εσείς θέλετε την ειρήνη που βασίζεται στο διάλογο. Πιστεύετε εσείς σε μια Ευρώπη η οποία δεν κάνει διαχωρισμούς ανάμεσα στην Ευρώπη του Βορρά και του Νότου, της Ανατολής και της Δύσης. Εσείς επίσης προέρχεστε από την, το κόμμα το οποίο κέρδισε τις εκλογές και είχε την προτίμηση των εκλογέων. Γιατί εμείς ε, συμμεριζόμαστε τη δική σας άποψη για το κράτος δικαίου ε, και γι' αυτό εμείς ε, βασιζόμαστε σε εσά για να υπερασπιστείτε και το κράτος δικαίου στην Ισπανία και την Ισπανική Ενότητα και ε, ε, εμείς είμαστε απέναντι σε αυτούς ε, που είναι κατά της Ευρώπης. Αυτοί που θα σας καταψηφίσουν είναι αυτοί που είναι κατά της Ευρώπης. Κυρία Φόντερ Λάγεν, εμείς και όλοι όσοι πιστεύουν στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σήμερα, πραγματικά σήμερα δεν πρέπει να αφήσουμε αυτήν την ευκαιρία να πάει χαμένη. Βασιζόμαστε σε εσά, αγαπητή κυρία. Ο κύριος Μωράης, δύο ε, κυρία κυρία Βαντελάιεν, υπάρχει λόγος για τον οποίο αναφερθήκατε διαδοχικά σε δύο από τα κρίσιμα θέματα, το οποίο η ομάδα μου ε, θεωρεί κύριε προτεραιότητε. Την επανεκκίνηση τη διαδικασία του Δουβλίνου και τη στήριξη ενό ενός ε, μηχανισμού για το κράτο δικαίου και παραθέτω τα λόγια σα. Ε, ο λόγο είναι ότι αυτά τα θέματα δεν είναι τα πιο σημαντικά. Αναφερθήκατε και στο θέμα του κλίματο, αλλά είναι θέματα που θα μπορούν να φέρουν την αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ξέρουμε αυτό και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποίησατε τι σωστέ λέξει, δώσατε τι επακεφαλίδε που θέλουμε να ακούσαμε, ε, αλλά όπως ακούσατε θα θέλουμε να έχουμε συγκεκριμένες ιδέες που κρύβονται κάτω από αυτά τα λόγια. Στη διαδικασία του Δουβλίνου, σε αυτό το σύμφωνο για την μετανάστευση, εσείς και εγώ γνωρίζουμε ότι απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία από τα κράτη-μέλη. Η αδράνεια του Συμβούλιο ε, έδειξε ότι δεν έγινε τίποτα στη μετανάστευση. Είδαμε κόσμο να πνίγεται στη Μεσόγειο. Υπάρχει αυτή η αδράνεια. Μπορείτε να κάνετε κάτι γι' αυτό. Αναφορθήκατε στα θέματα εξωτερικών σχέσεων, αλλά δεν το αναφέρετε εδώ. ποινικοποίηση τον ΜΚΟ, ε, η ανθρωπιστική διάδρομη, όλα αυτά είναι οι λεπτομέρειε που θέλουμε να ακούσουμε. Και στο θέμα τη στήριξη για το κράτο δικαίου. Και πάλι θέλουμε να δούμε τι λεπτομέρειε, το πολιτέ σχέδιο, τι κυρώσει στην Ουγγαρία και την Πολωνία. Κατονομάστε τι χώρε, γιατί αυτή είναι η ουσία. Ε, και πρόεδρε, θα μπορούσα να πω ε, ω ε, μέλο του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτή τη στιγμή γίνονται tweets ότι θέλετε παράταση, ό,τι και να γίνεται. Δεν είναι αυτό που είπατε. Σε μια επιστολή που αποστήλατε σε εμά, μα. το είπατε με εξωπρεπή τρόπο, μια παρά... αν χρειαστεί η παράταση για το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να υπάρχουν βάσιμοι λόγοι, καλοί λόγοι και ασχοληθήκατε με πραγματιστικό αξιοπρεπή στόχο ε, με το θέμα του Brexit. Είναι αυτή η εταιρική σχέση που θέλουμε να δούμε. Δεν θέλουμε ε, να ακούσουμε αυτά που ακούσουμε, ακούμε από άλλα μέλη αυτού του σώματος. Η πραγματιστική εταιρική σχέση είναι αυτό που θα μας πάει μπροστά. Ο κύριος Γκαρικάνο, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Βαντερλάινε, σας ε, συγχαίρω για την εξαίρετη ομιλία σας και την εξαίρετη συνεργασία που είχατε τις τελευταίες μέρες ε, με την ομάδα Renew Europe. Θέλω να πω στον, στους πράσινους ναι, ότι εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ε, αλλαγή σε σχέση με τις τελευταίες εβδομάδες. Νομίζω ότι εδώ ακριβώς υπάρχει αναγνώριση των διακυβευμάτων που αντιμετωπίζει, των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη απέναντι και σε αυτούς που θέλουν να αποτύχει η Ευρώπη, λαϊκιστές, εθνικιστές κλπ. Ναι, ε, θα πρέπει οπωσδήποτε οι ε, πολίτες να αισθάνονται αυτήν την ε, έννοια της προστασίας χωρίς όμως να υψώνονται τύχη γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προτείνουν αυτές τις ιδέες να υψώσουμε τύχη για να είμαστε ασφαλείς ξανά όχι. Η κυρία Φοντερ κατανοεί αυτούς τους προβληματισμούς και απέδειξε τον τελευταίο καιρό ότι μπορεί να δουλέψει μαζί μας για να οικοδομηθεί ακριβώς αυτή η Ευρώπη της δημοκρατίας, της συνένεσης ε, για το κλίμα, ε, για την ψηφιοποίηση για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λύνονται οι ευρωπαϊκές κρίσεις έχοντας στην πλάτη μας μια κακή επίλυση ευρωπαϊκής ε, κρίσης. Πιστεύω ότι και εμείς θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια και να πούμε ότι ίσως όλα δεν είναι εξαιρετικά αλλά ήρθε η στιγμή να είμαστε όλοι μαζί, να πούμε όχι στους εθνικισμούς, να πούμε όχι ε, στους ακραίους και να πούμε ναι στην κυρία Φόντερ Ο κύριος Ζαντό για ένα λεπτό παρακαλώ. Κυρία υποψήφια. Είπατε στις ακροάσεις ε, ότι, ότι υποστηρίζετε τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ. Ποια είναι η αξία όσον αφορά τις δεσμεύσεις για το κλίμα όμως, γιατί εδώ ε, σε αυτά τα πλαίσια υποστηρίζετε τον πρόεδρο Μπολσενάρο που πουλάει την ε, Αμαζονία στα μεγάλα συμφέροντα. Ποια είναι η δέσμευσή σας για ε, για τις γυναίκες όταν ο Μπολσενάρο καθημερινά επιτίθεται στις γυναίκες, ε, στους ομοφιλόφιλους, ε, στις δημόσιες αρχές. Δεν είναι αυτά, αυτές οι αρχές που εσείς υποτίθεται υπερασπίζεστε η υποστήριξη της Συμφωνίας Μερκοσούρ είναι η υποστήριξη της, των κακών τροφίμων, η υποστήριξη των μη δημοκρατικών αρχών. Εάν θέλετε εσείς να προωθήσετε ε, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, εάν θέλετε να μην πουλήσετε στις πολυεθνικές και στα λόμπινγκ ε, τις ευρωπαϊκές αρχές, ε, τότε να μην υποστηρίζετε την ακροδεξιά, να μην υποστηρίζετε την Βραζιλία και να μην υποστηρίζετε υποστηρίξετε και να σταματήσετε την συμφωνία Μερκοσούρ και να, να κοκκινήσετε το γραπτό και να το γυρίσετε πίσω όσον αφορά τη συμφωνία Μερκοσούρ. Mr. Madison, one minute. Uh, Ευχαριστώ, κύριε Φαντελάγεν. Θέλω ε, μόνο μερικές προτάσεις να πω. Πρώτα απ' όλα έχουμε πολύ συνέστημα και είναι κατανοητό διότι υπάρχουν, είναι μέρος της δημοκρατίας όλα αυτά. Συναντήθηκα με τον κύριο Τίμενες αρκετές φορές και ξέρω ότι είναι ένα από τα προβλήματα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, για την επιλογή του επόμενου υποψηφίου για την Κομισιόν αλλά ε, τι τις σχέσεις του, τις θέσεις του. Αν άκουγα την κυρία Φαντελάιν για το κλίμα, για την μετανάστευση, δεν υπάρχουν και πολλές διαφορές ανάμεσα στον κύριο Τίμερμανς και την κυρία Βόντερ Λάιεν. Είναι πραγματιστική πολιτική. Το κατανοώ αυτό, αλλά είναι γεγονός. Έχω μόνο 10, λεπτά, 10 ε, δευτερόλεπτα και θέλω να πω ότι όλα τα κράτη-μέλη στο χώρο Σέγγεν έχουν συμφωνήσει ότι θέλουμε να προστατεύσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα, όπως το κάνει η Ιταλία και η, το, η Ουγγαρία με το 1 δις ευρώ. Και θα πρέπει να σταματήσουμε την παράνομη διακίνηση ανθρώπων διότι ε, είναι σαν να δίνουμε εκατομμύρια στους διακινητές ε, και λέμε, ωραία, εμείς θέλουμε να ανοίξουμε τα σύνορα. Νομίζω δεν είναι έξυπνος τρόπος να προχωρήσουμε, αλλά καλή τύχη και ελπίζω να έχουμε και άλλους υποψήφιους. Ευχαριστώ. Mr. minute. Κύριος Επίνκ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Το πρώτο συμπέρασμα που εξάγω από όλα αυτά που ακούσαμε είναι ότι